take this Okay, friends, we'll start the voting session. Να ξεκινήσουμε, αγαπητοί φίλοι με τις ψηφοφορίες και έχουμε πολύ ωραίες ψηφοφορίες. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε επιθερχημένοι και αποτελεσματικοί. Αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε και τα μηχανήματα για να βλέπουμε τα αποτελέσματα. Να περάσουμε στην ψηφοφορία για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Αρφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Ποιος είναι υπέρ. Είναι ονομαστική ψηφοφορία. Έτσι λοιπόν θα την κάνουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Okay. Okay. Ah, it's too late. Okay, okay. The vote is closed. Λήξη. 44 υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές. Προχωρούμε στον επόμενο οργανισμό, στο ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. 45 υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές. Περνάμε τώρα στο Eurofound. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 43 υπέρ, 3 κατά, 3 εποχές. Περνάμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην επικοσμιοποίηση για την Αττική. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Και εγκρίνεται με 45 ψήφους υπέρ, 5 κατά και καμία αποχή. Προχωρούμε στην ε, έκθεση μπάλας. Το ίδιο. Και εδώ ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε έτσι ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Συμβαστική Α, άρχιτη ψηφορία. ψηφοφορία. Λήξη. Madam Harkin, did you have a question? No, just... Έχετε ερώτηση, κύριε Χαρκίν. Όχι, να πω ότι ξέχασα την κάρτα μου για τις ψηφοφορίες. Oh, um, Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Λήξη. 47 υπέρ, 2 κατά και καμία αποχή. Compromise M on... Συμβαστική M στη σελίδα 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 44 υπέρ, 6 κατά, Πάμε στην ε, τροπολογία 241 στη σελίδα 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 17 υπέρ, 33 κατά. Περνάμε στη συμβαστική C. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη για τη συμβιβαστική ΣΥ. Σαραντεφτά υπέρ. Καμία ψήφος κατά. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Βεβαίως και όχι λέει η πρόεδρος. 245 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και τη 245. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται με 47 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 246. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 43 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 247. Τμήμα 1. Είναι τμήματική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για το τμήμα 1. Πέρας. Εγκρίνεται. 28 ψήφους υπέρ, 23 κατά. Τμήμα 2. Γιατί 247. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται με 45 ψήφους κατά. Τροπολογία 248 καταπίπτει. Πάμε στη συμβαστική T. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Αναλλακτική συμβαστική τι όχι. Και πάμε στη σελίδα 17. Τροπολογία 285. Σελίδα 17. Άρχεται η ψηφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Με 26 ψήφους κατά. Τροπολογία 287. Άρχεται τη ψηφοφορία. And the vote is now closed. Λήξη. Απορρίπτεται. Με 27 ψήφους κατά. Συμβαστική S. Άρχεται ψηφορία. ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 292 μαζί με την τροπολογία 293. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνονται με 31 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται με 34 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 296. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται με 44 ψήφους κατά. Τροπολογία 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Λοιπόν, πάμε στη συμβαστική D. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται με 44 ψήφους υπέρ. Συμβαστική E. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται με 44 ψήφους υπέρ. Πάμε στη σελίδα 25. Τροπολογία 319. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται με 28 υπέρ. Τροπολογία 320. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται με 28 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 325. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 29 ψήφους κατά. Τροπολογία 326 μαζί με την 327. Άρχεται η ψηφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική G. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη εγκρίνεται. Συμβαστική H. Σε σελίδα 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται με 52 ψήφους υπέρ. Σελίδα 31. Πέτει 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Πέτει 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται με 37 ψήφους κατά. Τώρα ψηφίζουμε τη συμβαστική AO μαζί με τη συμβαστική BD. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται με 32 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική AP στη σελίδα 35. Άρχισε η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 41 ψήφους υπέρ. Περνάμε στην τροπολογία 382, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική AR. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται.

με 25 ψήφους υπέρ και 26 κατά. Σελίδα 39, συμβιβαστική AS, άρχεται ψηφορία. θα ψηφιστεί από κοινού με την συμβαστική BF αρχεται ψηφορία. Συμβαστική AS από κοινού την BF. Πέραση της Εγκρίνεται με 27 ψήφους. Ο κύριος Σούλτς, παρακαλώ. Ε, μια μικρή παράκληση θα χαιρόμασταν εάν ε, δεν λέγατε συνεχώς ποια σελίδα βρισκόμαστε διότι σε εμάς ε, είναι σε διαφορετικές σελίδες οπότε ε, δημιουργεί σύγχυση αυτό. Θα προσπαθήσω, δεν εγγυώμαι τίποτα, απαντάει η Πρόεδρος. Uh, now we are uh, on amendment 434. Uh, Περνάμε στην τροπολογία 434. Τροπολογία 434. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 46 ψήφους. Τροπολογία 435. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. απορρίπτεται. Τροπολογία 436 άρχεται. Ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Τροπολογία 438 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4.39». Πέρας της ψηφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 437. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 440. Ονομαστική ψηφορία. Άρχεται. Πέρας. απορρίπτεται. Τροπολογία 441, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 443, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. 444, αρχή της ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία. 445. Ονομαστική ψηφοφορία. Κυρία Πρόεδρε, ε, νομίζω ότι ε, χάσαμε μία ε, ψήφο στην 448. Όχι, απαντάει η πρόεδρος. Είμαστε στην τροπολογία 445. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Απορρίπτεται. 446 αποκινούμε την 447 άρχεται η ψηφορία πέρας εγκρίνεται με μία ψήφο παραπάνω 448 αρχή ψηφορία Όχι, συγγνώμη δεν ψηφίζουμε την 448. Πάμε στην 449 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 451 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 30 ψήφους. Τροπολογία 453. Άρχη της ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34. Άρχισε ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. 32. Άρχισε ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 42 ψήφους. Και περνάμε στην τροπολογία 456. Άρχη της ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 457. Άρχη της ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Άρχισε ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 29 ψήφους. Τροπολογία 458. Άρχισε ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική γιου. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 48 ψήφους. Και πάμε στην συμβιβαστική V. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 44 ψήφους. Τροπολογία 481. Αρχή του ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 29 ψήφους. Συμβιβαστική W. Αρχή του ψηφορία. Ψήφισε ένας παραπάνω από το EPP. Συμβαστική W. Πέρας της ψηφοφορίας. 49 υπέρ. 4 κατά. Πάμε στην συμβαστική AA. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 53 ψήφους τροπολογία. Πεντακόσια δεκατέσσερα, άρχισε ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική AB, άρχισε ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. στην τροπολογία 43 άρχεται τη ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται με 48 ψήφους συμβαστική AC Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Στην 37. Άρχεται η ψηφορία. 5.37 πέρας εγκρίνεται 5.38 πέρας της ψηφορίας εγκρίνεται 5.39 αρχής ψηφορία πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική AJ. Άρχιε ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 48 ψήφους. Περνάμε στην τροπολογία 562, άρχισε ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται μέσα από τα 5 ψήφους. Περνάμε στην τροπολογία 51, άρχεται ψηφορία. Πέρας. εγκρίνεται με 42 ψήφους. Τροπολογία 569, άρχης ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 570, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. Τροπολογία 571, άρχεται ψηφορία, πέρας, απορρίπτεται. 572 άρχισε ψηφορία πέρας απορρίπτεται. Τροπολογία 5.75 Άρχη συμφορία Πέρας Απορρίπτεται Περνάμε στην 5.79 Άρχη του συμφορία Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην AM 580. Άρχεται ψηφορία. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται με 52 ψήφους. Περνάμε στην τροπολογία 589. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 48 ψήφους. Περνάμε στην τροπολογία 54. Λέει η πρόεδρος. Συγγνώμη, 53 πρώτα. Τροπολογία 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 48 ψήφους. Και τώρα πάμε στην τροπολογία υπεριθμών 54. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. Συμβαστική I, Ι. Ψηφίζουμε. Για τη συμβαστική Ι. I. Πέρας. Εγκρίνεται. 46 ψήφοι πέρα. Συμβαστική K. K. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται με 48 ψήφους υπέρ. Συμβαστική J. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται με 45 ψήφους υπέρ. Ίσως και 46. Η 622 μαζί με την μαζί με την 623. Αυτές οι δύο. Και την 624 και 625. Υπέρ. Α, συγγνώμη. Ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 626 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 628 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 629. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 50 ψήφι πέρα. 630. Ψηφίζουμε. Πέρας. Πέντε ψήφοι υπέρ. Η 636 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 600 37 μαζί με την 638 και την 639. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 646. σαράντα Ψηφίζουμε. Πέρας. Συμβαστική L. Ζητήσετε το λόγο παρακαλώ. Όχι. Συμβαστική L. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 53 ψήφοι υπέρ. 649 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΤΑΦ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 51 ψήφι υπέρ. Συμβιβαστική AU. Ψηφίζουμε. Πέρας. Ψηφίζουμε την 657. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. Η 658 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 659. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 660. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 661. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. 28 η ψήφη υπέρ. Η 662 έναρξε και πέρας. Εγκρίνεται. Η 663. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 664. Η 666, λέει η πρόεδρος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 668. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται με 33 ψήφους υπέρ. Η 669 από κοινού με την 670. Έναρξε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 671 από κοινού με την 672. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 674. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 675. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 676 από κοινού την 677. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 678 αποκινούμε την 679. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 680 μαζί με την 681. Έναρξη ψηφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται.

Πέρας. Απορρίπτεται. Ή 683. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 59. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η εξήντα; Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 684. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 61. Υπέρ. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 685. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η 686 αποκινούμε την 687. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 542. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται με 41 ψήφους. Ή 688. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία υπαριθμών 689 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται η 690. Έναρξη. Πέρασε. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 694. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 695. Με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην τροπολογία περιθμών 1. Στη σελίδα 94 λέει η πρόεδρος. Την τροπολογία 1 λοιπόν ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 52 ψήφοι υπέρ. 62 τροπολογία υπέρ. Συγγνώμη, ψηφίσουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 52 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 2. Έναρξη. Καλησπέρα. 48 ψήφοι υπέρ. Σε μη βαστική Αλφα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται με 50 ψήφους υπέρ. 5-1 τη επιτροπή Αναφορών. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται οι δύο της Επιτροπής Αναφορών. Ψηφίζουμε. Πέρας. Πέτει 5-3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΒΒ. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Με 25 ψήφους υπέρ. 67. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 44 ψήφι 5-5. Έναρξη. Πέρας. 46 ψήφοι υπέρ. 5 4 ψηφιζουμε περας εγκρινεται 5 5 εναρξη περας 46 ψήφι υπερ 5 6. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 5-7. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 51 ψηφί υπέρ. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 76. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική βήτα. Έναρξη. Πέρας. 50 ψήφοι υπέρ. Τροπολογία 5. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 44 ψήφοι υπέρ. Τροπολογία 80 και 81. Ψηφοφορίες κατά τμήματα. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. Και είμαστε πάντα στην 81 πρώτο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα της 81, άρχιε της ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 82, έναρξη. λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 83. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 7. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τρομολογία 84. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική BC. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική BD. We go to compromise. Πάμε στη συμβαστική BE. Σελίδα 101. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 113. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 124. Συγγνώμη. Συμβιβαστική BG. Ψηφίζουμε αυτή τη συμβιβαστική BG, άρχεται ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 124. Άρχεται ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Άρχη ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 125. Έναρξη. Λήξη. Έχουμε ένα-δύο παραπάνω σοσιαλιστές. εγκρίθηκε. Τροπολογία 125, άρχιτη ψηφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική BH. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη για τη συμβαστική B έτσι εγκρίνεται με 51 ψήφους υπέρ. Πάμε στην τροπολογία 128, ονομαστική ψηφοφορία, Άρχιετη ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 129. Επίσης ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Απορρίφθηκε. Πάμε στην 130. Άρχεται η ψηφοφορία ονομαστική και εδώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Πέτει 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Α, όχι, εγκρίνεται. Πάμε στην πέτει 11. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική BI. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται με 46 ψήφους υπέρ. Πάμε στην 134 και εδώ ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Λήξη. Και απορρίπτεται. Τροπολογία 135. Άρχεται ψηφοφορία. Λήξη. Και εγκρίνεται με 48 υπέρ. Τροπολογία 136. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική BJ. Έναρξη. λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική BK, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 148, έναρξη. λήξη εγκρίνεται συμβαστική BL έναρξη λήξη εγκρίνεται με 43 ψήφους υπέρ 152 τροπολογία έναρξη λήξη Απορρίπτεται. Συμβεστική BM. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβεστική BN. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται με 37 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 153 λέει πρόεδρος. Καταπίπτει, συγγνώμη. Πάμε στην 154. Έναρξη. Λήξη. Υπήρχε τεχνικό πρόβλημα. Να ξαναψηφίσουμε. Ψηφίσαμε λοιπόν την 154 ελπίζω και απορρίφθηκε. Πάμε λοιπόν στην 155 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική BO. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική BP. Έναρξη. Λήξη. BQ έναρξη λήξη εγκρίνεται συμβαστική BR έναρξη λήξη εγκρίνεται Τροπολογία 173, έναρξη. Λήξη. Και απορρίπτεται. Πάμε στην 174, έναρξη. Λήξη. απορρίπτεται. Πάμε στην 175, έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβεστική BS. Έναρξη. Λήξη εγκρίνεται συμβαστική BT έναρξη λήξη εγκρίνεται με 52 υπέρ πάμε στην 5 17 έναρξη λήξη απορρίπτεται συμβεστική ποιού, Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 182. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Πάμε στην 187. Άρχεται η ψηφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 188. Έναρξη. λήξη. Έχετε όλοι ψηφίσει την 188. Ωραία, απορρίφθηκε. Συμβαστική BV. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. υπολογία Όχι, καταπίπτει. Πάμε στην 190, 191 και 518. Άρχεται η ψηφοφορία σε αυτές. Λήξη. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική BW, Έρχεται η ψηφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική BX, έναρξη. Λήξη. 195 υπέρ 8 κατά. Πάμε στην 196. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 198. Έναρξη. λήξει. Εγκρίνεται. 199. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 200. Έναρξη. Λήξη. εγκρίνεται 508 έναρξη λήξη εγκρίνεται 509 έναρξη λήξη απορρίπτεται 40 έναρξη λήξη εγκρίνεται και ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε Ψηφίσατε όλοι. Κλείνουμε λοιπόν την ψηφοφορία. yes. Then we vote on the... Ψηφίζουμε τώρα την απόφαση για έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 32 υπέρ, 17 κατά και 3 αποχές. Σας ευχαριστώ όλους. για αυτή την επίδειξη για το πώς ψηφίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.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 Ξεκινάμε την ε, ψηφοφορία για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Η ψηφοφορία για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα ξεκινήσει τώρα. shall what we should put it as well. Yeah, yeah, yeah, yeah. No, it's, uh, we vote. Mm. 47. We start by voting on amendment. Ξεκινάμε με την τροπολογία 47. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. 47 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας Απορρίπτεται. Περνάμε στην πρόταση της Επιτροπής. Ε, άρχεται ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε. Περνάμε στο ε, 1, τραν 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Για το υπόψη 1 τροπολογία τραν 2 απορρίφθηκε ε, τζούρι 2 άρχεται ψηφορία πέρας εγκρίνεται και περνάμε τώρα στα άρθρα κεφάλαιο 1, τροπολογία 257, υπέρ, κατά, Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 257. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στο άρθρο 1, τροπολογία 258. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστήκε 1. Άρχεται η ψηφορία. πέρας εγκρίνεται συμβιβαστική 2 άρχεται ψηφορία πέρας εγκρίνεται συμβιβαστική 6 άρχεται ψηφορία Πέρας. Εγκρίνεται με 42 ψήφους. Περνάμε στη γύρω 31, άρχη ψηφορία. Πέρας. απορρίπτεται. Τροπολογία 2.79, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. εγκρίνεται με 46 ψήφους. Πάμε στην Γιούρι 33, σε μένα είναι στη σελίδα 12, 13 λέει η πρόεδρος. Γιούρι 33, Αρχιετή ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τραν 28. Αρχιετή ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, περνάμε στην τροπολογία 30, 38, 338 πέρας απορρίπτεται περνάμε στην 33. πέρας απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβιβαστική 14. Ψηφίζουμε την συμβιβαστική 14. Αρχές ψηφοφορία. πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Πάμε στην σελίδα 30, λέει η πρόεδρος, όπου θα βρείτε τη συμβιβαστική 15, να έρχεται η ψηφορία. Πέρας. και εγκρίνεται με 46 ψήφους. Πάμε στην σελίδα 33. Τροπολογία 463. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην συμβιβαστική 16. Άρχεται η ψηφορία. Συμβιβαστική 16. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται με 48 ψήφους. Ψηφίζουμε για την συμβιβαστική 17. Πέρας. Εγκρίνεται με 46 ψήφους. Συνεχίζουμε στην τροπολογία 475, άρχεται ψηφορία. πέρας απορρίπτεται κατά δύο ψήφους περνάμε στην συμβιβαστική 18 άρχης ψηφορία πέρας εγκρίνεται με 49 ψήφους περνάμε στην budget 12 σελίδα 36 το πρόεδρος άρχισε ψηφορία, πέρας απορρίπτεται συμβιβαστική 19 άρχισε η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται με 47 ψήφους Συμβαστική 20. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 48 ψήφους. Περνάμε στη συμβαστική 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 47 ψήφους. Περνάμε στην τροπολογία 504, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 27 ψήφους. 505, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. budget 13 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται με 30 ψήφους περνάμε στη Γιούρη 46 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται Περνάμε στην τροπολογία 506. Αποσύρθηκε, οπότε περνάμε στην 507, αποκινούμε την 508. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 29 ψήφους. ψηφίσουμε την 509 από κοινού με την 510, 511 και Γιούρι 46. Άρχιε ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 45 ψήφους, συμβιβαστική 22, άρχιε ψηφορία. Πέρας. εγκρίνεται με 46 ψήφους. Περνάμε στη συμβιβαστική 23, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 50 ψήφους υπέρ, μία κατά. Συμβαστική 24, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 45 ψήφους. Περνάμε στην τροπολογία 528, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται Περνάμε στην 529. Όχι, Γιούρι 46. Ψηφίσουμε για τη Γιούρι 46. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 530. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας απορρίπτεται. Δεν θα ψηφίσουμε την 531, οπότε περνάμε στην 532. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίσουμε την 533, άρχεται η ψηφορία. Πέρας απορρίπτεται. Περνάμε στην 534, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην συμβιβαστική 25. Πέρας της ψηφορίας εγκρίνεται. Πηγαίνουμε τώρα στη σελίδα 50. Συμβαστική 28. Άρχιτσι Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε στην συμβιβαστική 29, άρχιτη ψηφοφορία, πέρας. 45 ψήφοι υπέρ και μία κατά. Περνάμε σε ψηφοφορία κατά τμήματα για την τροπολογία 603, το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 29α. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. και εγκρίνεται. Συμβαστική 30. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 46 ψήφους. Περνάμε στην τροπολογία 612. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας απορρίπτεται. Συμβιβαστική 31. Αρχή ψηφοφορία. ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 32. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 43 ψήφοι υπέρ. Συμβαστική 33. Στη σελίδα 58. Λέει πρόεδρος, ψηφίζουμε. Πέρας. 46 ψήφοι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 34. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται με 48 ψήφους υπέρ. Οι 650. ψεφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Γιούρι 49 της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Η 49. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 651. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 655. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 656. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 35. Έναρξη. Πέρας για τη συμβαστική 35 εγκρίνεται με 42 ψήφους υπέρ. Γιούρι 50. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 667. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 668. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 669. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 355 55. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε τώρα την 670. Έναρξη. Πέρας. 671. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 672. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 673. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 674. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Γιούρι 50. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Της Επιτροπής Μεταφορών η παριθμών 56. Ψηφίζουμε. Τραν 56. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 675 μαζί με την Γιούρι 50 από κοινού. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 36. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Γιούρι 50. Έναρξη. Ο κ. Λέναρτς. Ένα τεχνικό σημείο να επισημάνω, γιατί νομίζω ότι στην συμβαστική 36 ψηφίσαμε με τη Γιούρι 50 γιατί είναι ταυτόσημη με την 651. Είναι το σημείο που αντιστοιχεί στην παράγραφο 4, λέει η Πρόεδρος. Γι' αυτό το ψηφίζουμε. Αν ψηφίσετε όλοι για την γύρι 50, πέρας. Και απορρίπτεται. 680. Την 679, διορθώνει πρόεδρο. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 680. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. ΦΑΜ 34. Έναρξη. ΦΑΜ 34. Έναρξη και πέρας. Απορρίπτεται. Η 681 και η Γιούρι 51 και ψηφίζουμε παρακαλώ. 38 ψήφι κατά. Απορρίπτεται. 52. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 682. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 67. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ. Και περνάμε στην 690. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 691 αποκινούμε την 360. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τραν 61. Έναρξη. Και πέρας. Απορρίπτεται. Η 692 αποκινούμε την Γιούρι 51. Η 692 από κοινού με την Γιούρη 51. Έναξε. Πέρασε. Τραμ 62 τώρα. Συγγνώμη, μόνο την τραν 62 ψηφίζουμε. Την τραν 62. Έναρξη. And the vote is now. Και περασε Απορρίπτεται. Σχόλια εκτός μικροφώνου από την αίθουσα. The result of το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την 692. 9 uh, ψήφοι υπέρ και 36 κατά. Μην τα αποχιάσει. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Και τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία του κυρίου Κώσα υπαριθμών 693. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. ΦΑΜ 32. 35, συγγνώμη. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 694. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται.

Πέρας. 39 οι κατά, 10 οι υπέρ. Απορρίπτεται. Ή 697. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τραν 63. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Γιούρι 51. Αποκινούμε την 698. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Γιούρι 51. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ. Άρθρο 13. Δεν ψηφίζεται. Άρα περνάμε στην συμβαστική υπέρθμονη 37. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 43 ψήφοι υπέρ. Συμβιβαστική υπαριθμό 38. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 40 ψήφοι υπέρ. Συμβιβαστική 39. Έναρξη. Πέρας. Σαράντα πέντε ψήφοι υπέρ εγκρίνεται. Συμβιβαστική σαράντα. Έναρξη. Και πέρας. Σαράντα πέντε ψήφοι υπέρ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 41. Έναρξη. Πέρας. Για την 41 εγκρίνεται 46 ψήφοι υπέρ. Συμβαστική 42. Έναρξη. Πέρας. 47 ψήφοι υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 754. Έναρξε. Και πέρασε. 43 ψήφοι πέρα εγκρίνεται. Και περνάμε στη Γιούρη 52. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται με 44 ψήφους. Γιούρη 52. Ψηφίζουμε. και πέρας. Απορρίπτεται με 42 ψήφους. Έχουμε την 754. Έναρξη. Και πέρας. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 43. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται με 44 ψήφους. Η 769 έναρξη. Και πέρασε. Απορρίπτεται. Η 770 παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 771. Από κοινού με την Γιούρι 54. Έναρξη. Και πέρασε. Απορρίπτεται με 45 ψήφους. Συμβαστική 44. Έναρξη. Και πέρασε. Εγκρίνεται με 43 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 778. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 779. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 780. Αποκινούμε την Γιούρι 55. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Λίμπε 46. Έναρξη. Και πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 781 από κοινού με την 858. Τις ψηφίζουμε από κοινού παρακαλώ, έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην συμβαστική 45. Έναρξη. Πέρας. 43 ψήφοι υπέρ. Στην 795 ψηφίζουμε τώρα. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 45α. Έναρξη. Πέρας εγκρίνεται με 47 ψήφου υπέρ. Περνάμε στη συμβαστική 46, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται με 39 ψήφου υπέρ. Yes. We go to compromise 47. Συμβαστική 47, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται με 40 υπέρ. Τροπολογία 822. Σελίδα 84 λέει πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική 48. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Με 46 ψήφους Πάμε Στιφάν 38 έναρξη Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 831. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται με 42 ψήφους. Πάμε στη Λίμπε 49. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Γιούρι 58. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 830. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται με 45 ψήφους. Τροπολογία 834. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται με 45 ψήφους υπέρ. Πάμε στην 836 με τη Γιούρι 62 μαζί. Είναι συμβατές. Ψηφίζουμε την 836 μαζί με την Γιούρη 62, έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 838. Άρχεται η ψηφοφορία. να Απορρίπτεται. 839. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 842. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείξε. Σαράντα υπέρ, οκτώ κατά. Συμβαστική σαράντα εννιά. Έναρξη. 46 υπέρ. And the vote is... Πάμε στην επόμενη τροπολογία, 852. Έναρξη, λήξη. Εγκρίνεται. Πάμε στην 855. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 269. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 856 μαζί με τη Γιούρη 70. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Πάμε στην 857. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική 49α. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 50. Άρχεται η ψηφοφορία. λήξη 52 υπέρ πάμε στη συμβαστική 51 έναρξη λήξη εγκρίνεται με 48 υπέρ πάμε στη συμβαστική 52 έναρξη λήξη Εγκρίνεται με 47 ψήφους υπέρ. Πάμε στην τροπολογία 897. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Πάμε στη Γιούρι 73. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Πάμε στην 898. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Με δύο ψήφους. 899. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. ΦΑΜ 42. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 900. Έναρξη. Λήξη απορρίπτεται πάμε στην τροπολογία 901 έναρξη λήξη εγκρίνεται με 46 ψήφους πάμε στην 902 έναρξη λήξη Εγκρίνεται με 45 ψήφους. 923. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Εννιακόσια πέντε. Καταπίπτει ή 904. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ. Εδώ πέρα αναφέρεται ότι η 903 δεν θα ψηφιστεί αν εγκριθεί ο συμβιβασμός 50 και πριν από λίγο ψηφίσαμε και άλλη μια τροπολογία όπου και πάλι αναφερόταν ότι κανονικά θα πρέπει να καταρπέσει εφόσον ε, εγκρίνεται η συμβαστική 50. Άρα η 904 θα την ψηφίσουμε ναι ή όχι, δεν το έχω καταλάβει καλά. Yes, well, ε, ε, η 904 καταπίπτει, καθώς υιοθετήσαμε τη συμβαστική 50. Αυτός είναι ο λόγος. Ναι, αλλά η Γιούρι 62 και η τροπολογία 836 τις ψηφίσαμε επίσης. Παρά το γεγονό ότι αναφέρεται από δίπλα ότι θα έπρεπε να καταπέσουν αν περάσει η συμβιβαστική 50. Αυτές λοιπόν τις δύο τις ψηφίσαμε complicated if you... an article which is not mm-hmm. you If it, I mean, if I understand correctly, the previous... Αν κατάλαβα καλά, η προηγούμενη ψήφος ε, που αφορούσε τη συμβαστική 50 έλεγε ότι θα καταπέσει, αλλά εμείς κατόπιν αιτήματος των πρασίνων αποφασίσαμε να το ψηφίσουμε ξεχωριστά. Όμως αυτή εδώ η τροπολογία, η 904, Όντως καταπίπτει και δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Σωστά, μάλιστα. Το λύσαμε λοιπόν. Λοιπόν, καταλάβαμε γιατί συνέβη αυτό και πάμε στην τροπολογία 905 που θα ψηφιστεί μαζί με τη Γιούρι 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Πάμε στην ε, FAM 43. Την budget 18. Συγγνώμη. Θα πρέπει να ψηφίσουμε την budget 18. Άρχεται η ψηφοφορία λήξη. Και πάμε στη ΦΑΜ 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Πάμε στην 906. And the vote is closed. Λήξη. Και εγκρίνεται με 42 υπέρ. Budget 19. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ. Γιούρι 75. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται με μία παραπάνω ψήφο υπέρ. Πάμε στη ΦΑΜ 44, έναρξη. Λήξη. Και απορρίπτεται με μία ψήφο. Κατά παραπάνω. Πάμε στην 907 και στην 908 μαζί. Έναρξη. Λήξη. Πάμε στη Γιούρι 76. Όχι, συγγνώμη. Πρέπει να ψήσουμε την 908. Ψηφίζεται για την 908. Λήξη απορρίπτεται. Γιούρι 76, έναρξη, λήξη, εγκρίνεται. 909, έναρξη, λήξη, εγκρίνεται. Συμβαστική 55, πρόεδρε, συγγνώμη, Μπορείτε να μας αφήσετε χρόνο να ψηφίσουμε. Κάποια δευτερόλεπτα παραπάνω για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ένα-δύο δευτερόλεπτα ακόμα. Ευχαριστώ. Βεβαίως. Είναι μια έκτακτη συνεδρίαση ψηφοφοριών με ώρες και ώρες ψηφοφοριών. θα επιβραδύνουμε αν σας διευκολύνει. Η πλειοψηφία θέλει να πάμε πιο γρήγορα. Λοιπόν, πάμε στη συμβαστική 55. Έναρξη. Λήξη. Είχαμε 45 υπέρ, 3 κατά. Πάμε. Στη συμβεστική 56. Έναρξη. Λήξη. 48 υπέρ, ένας κατά. Πάμε στην τροπολογία 922. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Πάμε στην 923. Έναρξη. Λήξη για την 923. Απορρίπτεται με 44 ψήφους. Πάμε στη συμβαστική 57. Έναρξη. Λήξη. υπέρ. Πάμε στη Λίμπε 52. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 26 ψήφους κατά. Περνάμε στην 926 μαζί με τη Γιούρη 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται με τρεις ψήφους. Πάμε στη ΛΥΜΠΕ 53 μαζί με την budget. Α, συγγνώμη. Δεν είναι μαζί οι τροπολογίες αυτές. Περνάμε στη ΛΥΜΠΕ 53. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Budget 21. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Άρθρο 38. Λίμπε 54 και Γιούρι 79 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Γιούρι 80. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική 58. Έναρξη. Λήξη και εγκρίνεται με 43 ψήφους υπέρ. Go to... Ε, Περνάμε στην τροπολογία 932. Αποκινούμε την Γιούρι 81. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 933 Αποκινούμε την Yuri 82 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται με μία ψήφο παραπάνω άρθρο 43 τροπολογία 934 άρχεται η ψηφοφορία πέρας Απορρίπτεται. Τροπολογία 935. Ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 936. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εκκρίνεται με 41 ψήφους. Λίμπε 55. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Γιούρι 83. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 43 ψήφους. Συμβαστική 59. Αρχίζει ψηφορία. Πέρας. Σαράντα πέντε υπέρ, τέσσερις κατά. και περνάμε στην σελίδα 150, 105 συμβαστική 64 υπέρ κατά θα ψηφίσουμε λοιπόν Σαρδα υπέρ συμβαστική ψηφίσουμε από κοινού τις συμβιβαστικές 61, 62 και 63. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. 44 υπέρ. Περνάμε στις ιδεολογικές σκέψεις. Συλλογική σκέψη 1, τροπολογία 54, 55, γιουρι όχι. Μόνο την τροπολογία 54. Αιτιολογική σκέψη 1 λοιπόν, ε, τροπολογία 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Γιούρι 3. Πέρας. Απορρίπτεται. Λιμπένα. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην, στην ε, θεολογική σκέψη 2, τροπολογία 56, αρχίζει η ψηφορία, πέρας, απορρίπτεται, 57, αρχίζει η ψηφορία, πέρας, απορρίπτεται, Περνάμε στην τραν 3. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. και απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Περνάμε στην τροπολογία 59, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Λίμπε 2 και Γιούρι 4 από κοινού ψηφοφορία ταυτόσιμες Άρχη ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 42 ψήφους. Περνάμε στην Λίμπε 3. Άρχη ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 29 ψήφους. Περνάμε στη Λίμπε 5. Πέρας της ψηφορίας εγκρίνεται με 37 ψήφους. Αιτιολογική σκέψη 3. Τροπολογία 60. αρχή της ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 61. αρχή ψηφοφορία. ψηφορία πέρας απορρίπτεται Λίμπε 7 και Γιούρι 5 από κοινού άρχεται η ψηφορία πέρας απορρίπτεται 27 ψήφους Λίμπε 8 άρχεται η ψηφορία πέρας 40 υπέρ 7 κατά ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 62 άρχιες ψηφορία πέρας απορρίπτεται με 27 ψήφους τροπολογία 63 η ψηφορία Πέρας. Απορρίπτεται με 27 ψήφους. Τροπολογία 1. Του κυρίου Λένας άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται με 37 ψήφους. Αιτιολογική σκέψη 4B, 4B, άρχεται η ψηφοφορία και την τροπολογία 64. Πέρας. Απορρίπτεται. Λίμπε 6. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 65. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 66, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 67, άρχεται ψηφοφορία. Συγγνώμη. Η 67 καταπίπτει. Το ίδιο συμβαίνει και με την ΛΥΜΠΕ 4, οπότε πηγαίνουμε κατευθείαν στην συμβαστική 4. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται με 37 ψήφους υπέρ, 5 κατά. Και περνάμε στην τροπολογία 86. αρχίζει η ψηφορία Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην Τροπολογία υπαριθμών 4. αρχιετή ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβιβαστική 5. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Ε, εγκρίνεται με 46 ψήφους υπέρ. Περνάμε στην τροπολογία 101. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 39 ψήφους. Τροπολογία 102. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας απορρίπτεται ή budget ενα άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται κατά μία ψήφο παραπάνω λίμπε 11 προφορική τροπολογία από το S&D Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 44 ψήφους. Περνάμε τώρα στην συμβιβαστική 14α. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 42 ψήφους. Περνάμε τώρα στην Τροπολογία 114. άρχιε η ψηφορία, Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 115. άρχιε η ψηφορία, Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην Χιούρι 9. Άρχεται η ψηφόρία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην Συμβαστική. 60. Άρχεται ψηφορία. ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 38 ψήφους. Περνάμε στην λίμπη 14, αρχή ψηφορία. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 128. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 36 ψήφους. Περνάμε στην τροπολογία 7, άρχια της ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 38 ψήφους. Περνάμε στην Γιούρι 10, τη ψηφοφορία. πέρας απορρίπτεται τροπολογία 132 άρχεται ψηφορία πέρας απορρίπτεται λίμπε 15 Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην συμβιβαστική 14 β. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε στην Τροπολογία 142. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε στην συμβιβαστική 15α. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας και εγκρίνεται με 46 ψήφους. Περνάμε στην τροπολογία 157. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 158. πενήντα οκτώ. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Επίσης απορρίπτεται. Οπότε συνεχίζουμε στην 159. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην Yuri 13. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται συνεχίζουμε στην 160 άρχιζε η ψηφορία πέρας απορρίπτεται Ψηφίσουμε τώρα για την 162, αρχίσει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πηγαίνουμε στην 163 τώρα. Από κοινού με την ΛΥΜΠΕ 16, μια και είναι ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας απορρίπτεται τραν 10 άρχεται η ψηφορία πέρας απορρίπτεται οπότε περνάμε στην αιτιολογική σκέψη 14 και τη συμβεβαστική 26 άρχεται η ψηφορία πέρας και εγκρίνεται με 44 ψήφους. Περνάμε στην τροπολογία 173, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Σχόλιο εκτός μικροφώνου από την αίθουσα. Σελίδα 123 σε μένα, λέει η Πρόεδρος, τροπολογία 173. Θα δω τέτοιου εφιάλτες, λέει ο Πρόεδρος. Βρήκατε την ε, τροπολογία 173, μπορούμε να ξαναψηφίσουμε. Oh, Προχωράμε. Ξέρετε όμως ότι τώρα περνάμε πλέον στη συμβαστική 36α. 36α ψηφίζουμε. Έναρξη της ψηφοφορίας. 44 είναι η ψήφη πέρα Αιτιολογική σκέψη 16. Η τροπολογία 181. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 182 συμβατή με την 181, ίσως και να πρέπει να τις έχουμε ψηφίσει μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει ψηφίσουμε την 182. Την ψηφίζουμε. Την 182, παρακαλώ ψηφίζουμε. If there are protesters, but Amendment 182 182 ψηφίζουμε. Τραν 13 ψηφίζουμε. Έχουμε ξεκινήσει την ψηφοφορία για την Τραν 13. Πέρασε. Απορρίπτεται. ΦΑΜ 6. Έναρξη. Πέρας. Για την φάμα 6. Απορρίπτεται. Η 42α. Έναρξη. Πέρας. 38 ψήφοι υπέρ, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 43α. Έναρξη. Πέρας για τη 43α. 45 ψηφί υπέρ, μία κατά. Τροπολογία 201. Αλλαξή ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 53. Πέρας. 41 ψήφη υπέρ. Αιτιολογική σκέψη 22, η 210 τροπολογία. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 34 ψήφοι κατά. 211 τροπολογία. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 54. We vote on compromise 54. Συμβαστική 54. Πέρας. Εγκρίνεται με 45 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 218 από κενού με την 219. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται με 32 ψήφους. Η τρία της Επιτροπής Προπολογισμού. Budget τρία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 220. Εντάξει. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τραν 17. Έναρξη. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η 221. έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Γιούρι 20. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Η λίμπη 22. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 25α και η 222 τροπολογία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Budget 4. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 59α. Έναρξη. Πέρας. Έγκριση με 36 ψήφους. Υπέρ. Συμβιβαστική 44α. Έναρξε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 229. Έναρξη. Και πέρασε. Απορρίπτεται. 8. Έναρξη. Πέρες. Απορρίπτεται. ΦΑΜ 9. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 65. Έναρξη. Και πέρασε. Εγκρίνεται. Στην 241 πάμε τώρα, στην σελίδα 133. 241 της κυρίας Μαραμπιζότο. Έναρξη. Και πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 244. Έναρξη για την 244. Πέρας. Απορρίπτεται. Διακόσια σαράντα εννέα. Έναρξη. 249. Τέρι Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Φαμ 10. Έναρξη. Και πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 27. Έναρξη. Πέρας εγκρίνεται με 43 ψήφους. Συμβιβαστική 66. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 39 ψήφοι υπέρ. Περνάμε τώρα Συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Εντελογική σκέψη 37 και Γιούρι 25 παρακαλώ. Ένταξη ψηφοφορία. Και πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 256. Τεριρέντκε. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Λίμπε 26. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα είναι 33 ψήφοι υπέρ, μία εξικατά. Και σας ευχαριστούμε. έχουμε να ψηφίσουμε και την απόφαση για την έναρξη των ε, διαθεσμικών ε, διαπραγματεύσεων. Πάμε λοιπόν. Όσοι είναι υπέρ λοιπόν της έναρξης των διαπραγματεύσεων. 33 λοιπόν ε, υπέρ, 9 κατά. Και 6 αποχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαραθώνιος πραγματικά η σημερινή ψηφοφορία. Έχουμε και άλλες ψηφοφορίες όμως. Okay, shall we say five minutes... Να κάνουμε ένα του διάλειμμα αν θέλετε. Πέντε λεπτάκια. Πέντε λεπτάκια σας δίνω.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 Okay, friends, uh, we have done... Λοιπόν, έχουμε κάνει την περισσότερη δουλειά. αλλά έχουμε ακόμα 30 λεπτά, αν είμαστε αποτελεσματικοί. Gather here and put ourselves together. Για να προσπαθήσουμε να συγκεντρωθούμε she wanted now. Yeah, yeah. Hmm? Very, very Minority opinion. Okay, I'll give the floor to Madame Melan. Να δώσω το λόγο στην κυρία Ελάν που έχει, το έχει ζητήσει. Ναι, ευχαριστώ. Σας ε, ευχαριστούμε. Πήραμε μια να, να εκφράσω την ε, ε, Μια ψηφική άποψη, η γαλλική αντιπροσωπεία του ΕΝΕΦ ε, δεν είναι αλληλέγγυη με το έργο που έγινε στο φάκελο αυτό για πολλούς λόγους, γιατί προβλέπεται για να ανακουφίσει την ε, ανεπάρκεια την ανικανότητα της ίδιας της Κομισιόν. Έτσι, λοιπόν, ε, υπάρχει, ε, αυτός, ο αυτός ο συγκεντρωτισμός ε, δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει ο οργανισμός και σίγουρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το αμφισβητήσουμε. Έτσι λοιπόν ο οργανισμός αυτός έτσι όπως δημιουργείται δεν έχει τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που της τίθενται. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω στον συνάδελφο από την ΕΝΕΦ ότι αν είχε αυτέ τι ανησυχίε, θα ήταν καλό αν είχε εμφανιστεί έστω και μία φορά στη συνάντηση των σκιωδών όταν τα συζητούσαμε όλα αυτά. Okay, uh, then we proceed with the voting. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Έχετε Το είναι έκθεση για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες ενωπιών σας. Θα ξεκινήσουμε με τη συμβαστική 11. Με ένα τεσχυρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 14. Υπέρ. Against. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην βαστική τρία Σελίδα τρία Στο δικό μου έγγραφο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε τη συμβαστική τρία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμβιβαστική 3. 39 υπέρ, 3 κατά. Να πάμε στη συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχέ συγκρίνεται πάμε στη συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στη συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Γιούρι 2 και 3 καταπίπτουν. Ψηφίζουμε την τροπολογία 29 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται. Με στην τροπολογία 35 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 39. Λήξη. για την 39 25 υπέρ 16 κατά Πάμε στη συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας 4 τροπολογία γιούρι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 47. Περ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Τροπολογία 63. Υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ κατά να ελέγξουμε την τροπολογία 11 What was the result? 20. 21 κατά, 14 υπέρ. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για 15 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι εγκρίνεται Γιούρι 14 Τροπολογία 74 υπέρ. Κατά. Εποχές. Πρέπει να ελέγξουμε την 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Κατά μία ψήφο. 75 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται γύρω 15 καταπίπτει πάμε στην τροπολογία 17 υπέρ κατά εποχέ. ελέγχουμε τη 17 Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε το σχέδιο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται με 43 ψήφους υπέρ. Και καμία ψήφο κατά. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια. Θα ψηφίσουμε και την απόφαση για την έναρξη των ε, διοργανικών διαπραγματεύσεων, όπως προτείνεται από την εισηγήτρια. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια για την ε, πολλή δουλειά που είναι και πολύ σημαντική. Τώρα, θα ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης που θεσπίζει το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και τις αξίες. Ξεκινάμε την τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται θα έλεγα. Να ελέγξουμε τον τίτλο. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Προχωράμε στην τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Συμβεστική 11 υπέρ. Κατά εποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά εποχές Πρέπει να ελέγξουμε την 12. Δεν είναι σαφές. Λήξη. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να σηκώνετε τα χέρια σας, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. 32 υπέρ. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. εποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 97 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε την 102 άρχεται η ψηφοφορία λήξη απορρίφθηκε η 102 πάμε στην 103 υπέρ κατά Αποχές ελέγχουμε την 103. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Και προχωράμε στην 104 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβεστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. προφορική τροπολογία από την εισηγήτρια υπέρ κατά εποχές πρέπει να ελέγξουμε την 106 άρχεται η ψηφοφορία λήξη απορρίπτεται 22 ψήφους κατά Πάμε στην τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Εποχές. Να ελέγξουμε τη 16. Έναρξη. Λήξη. Τρίτα τρεις κατά απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε την 108 έρχεται η ψηφοφορία έρες Γκρίνεται. Στην 28 πάμε, υπέρ, κατά, εποχές, να ελέγξουμε την 28. Άρχεται ψηφοφορία, λήξη, εγκρίνεται. Με 35 ψήφους υπέρ. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Υπάρχουν ε, κάποιες ψηφοφορίες όπου οι συνάδελφοι δεν σηκώνουν όλοι το χέρι, αλλά βλέπουμε το συντονιστή κάθε ομάδας ε, και όταν ε, οι συντονιστές των κύριων ομάδων, των βασικών ομάδων, κάνουν το ακόλουθο σημάδι, δίνουν το ακόλουθο μήνυμα, Νομίζω δεν χρειάζεται πάντοτε να ελέγχουμε, γιατί κάθε φορά που χάρη που το ΕΛΚ ε, σηκώνει το χέρι προς τη μία την άλλη κατεύθυνση, έχουμε 33 ψήφους ε, κτλ. Well, I'm grateful if you raise your hand. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θα σας παρακαλούσα να σηκώνετε τα χέρια σας, ε, καθώς έχουμε ήδη ψηφίσει για ώρες και είμαστε όλοι κουρασμένοι. Αλλά ας τελειώσουμε και αυτές τις διαγνωμοδοτήσεις. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά εποχέ, συγκρίνεται 31 υπέρ κατά εποχέ, συγκρίνεται 32 υπέρ κατά εποχέ, συγκρίνεται 33 υπέρ κατά εποχέ. εγκρίνεται ή να ελέγξουμε, να ελέγξουμε τη 33 Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 λέει πρόεδρος. Συγγνώμη. 36 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχέ συγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά εποχέ, συγκρίνεται. Συμβαστική όχι. 54 υπέρ κατά εποχέ, απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας 15. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 αυτή είναι συμβατή με την 9 υπέρ για την 74 κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές υπολείπτεται 76 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 80 όχι 78 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 80 And the vote is closed. Λήξη. Γκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της γνωματότησης όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Και το αποτελεσμα είναι 38 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και μία αποχή. Και σας ευχαριστώ για αυτή την τρομερή μέρα. Ε this, this so shall we vote on this? We have one vote left. No presentation. Presentation. No, sorry, we have a Έχουμε μια παρουσίαση. Και είμαι σίγουρη ότι πολλοί θα μείνετε για να ακούσετε την παρουσίαση αυτή. Ε, ε, to be polite, ε, since, we... Και για να είμαι ευγενική, Έχουμε καλέσει Αντρέα Μπρότελ που είναι project leader και ερευνήτρια και θα μας πει θα μας μιλήσει για το θέμα της άμβλησης του διασμού στην αγορά εργασίας. Ένα από τα κύρια θέματα για μας ε, στην Επιτροπή αυτή. Αν μπορείτε να περιμένετε ένα λεπτό για να ηρεμήσουν οι συνάδελφοι, πιθανόν θα μείνουν και θα σα ακούσουν. And if you are not planning to Και αν δεν σκοπεύετε να μείνετε και να ακούσετε την προσκεκλημένη ομιλήτρια, παρακαλώ αποχωρήστε από την αίθουσα ησύχω. Ευχαριστώ και έχετε το λόγο. Okay, thank you very much. And... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να έρθω να μιλήσω εδώ. Χαίρομαι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους αποφάσισαν να μείνουν. Κατανοώ ότι ήταν δύσκολη η μέρα. Θα παρουσιάσω εντάχει τα αποτελέσματα μιας έρευνας ε, που μας ε, ζητήθηκε να κάνουμε εκ μέρους της Επιτροπής ε, Απασχόλησης, εκ μέρους της οργάνωσης ECORIS. Βρισκόμαστε στην Γερμανία σχετικά με τον διεισμό της αγοράς της εργασίας και τι κάνουν τα κράτη-μέλη για να το καταπολεμήσουν. Θα ήθελα να παρουσιάσω εντάχει τα αποτελέσματα. Ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να επικεντρωθούμε πάνω σε αυτό είναι ε, διότι ε, η ε, προσωρινή απασχόληση αυξάνεται τα τελευταία χρόνια η προσωρινή απασχόληση αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των αγορών εργασία ε, στην Ευρώπη κατά μέσο όρο στο 12% ενώ σε κάποιε χώρε όπως είναι η κατοχώρηση η Ισπανία η Πορτογαλία, η Πολωνία είναι στο 15% και το πώς επηρεάζει ε, τους ανθρώπους θεωρούμε ότι είναι υψηλότερη ανάμεσα ε, στους νέους, στους χαμηλότερα καταρτισμένους, στους μετανάστες καθώς επίσης και σε, στον τομέα παροχής υπηρεσιών για άτομα που έχουν χαμηλότερη κατάρτιση. Και αν δείτε εδώ τα διάφορα κράτη-μέλη, η κόκκινη γραμμή είναι στο 12% αφορά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ε, μετρήσαμε δύο περιόδους, το 2006 και το 2016, για να δούμε την προσωρινή απασχόληση σε σχέση με την ολική απασχόληση και συνολικά βλέπουμε ότι αυξήθηκε σε 18 χώρες, μειώθηκε σε 8 συνολικά, οπότε βλέπουμε μια οδυνατική τάση στις περισσότερες χώρες. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή λίγο πολύ παρέμεινε ο ίδιος. Τώρα όσον αφορά τους ε, βασικούς ε, δείκτες είναι ένα πολύπλοκο ε, στοιχείο. Βρήκαμε όμως ότι οι εργαζόμενοι προτιμούν να αποδεχτούν τέτοια συμβόλαια σε περίπτωση που δεν έχουν μόνιμη θέση εργασίας. Ο ρόλος της εθνικής νομοθεσίας και των εθνικών θεσμών παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, ενιαία σύμβαση ορίστου ε, χρόνου. Ε, έχουμε εκπαιδευτικά συστήματα σε χώρες όπως είναι η Αυστρία, Δανία και η Γερμανία όπου έχουμε μαθητείες κομμάτι της αγοράς εργασίας. Τώρα όσον αφορά επισφάλεια βλέπουμε ότι ε, έχουν χαμηλότερους μισθούς, δεν έχουν εκπροσώπηση στα σωματεία, έχουν περιορισμένες δυνατότητες ε, στην ε, ανέλυξη την καριέρα τους, στην εκπαίδευση, το οποίο δυσχεραίνει την επισφάλεια. Με αποτέλεσμα πολλοί να μένουν κολλημένοι σε τέτοιο πλαίσιο εργασίας ή αν μπορούν να ε, βελτιώσουν τις ε, συνθήκες. Ε, εδώ βλέπουμε ανηλικιακή ομάδα πως έχει η κατάσταση ηλικιακη ομαδα πως εχει η κατασταση σχετικα με την περίοδο 2006-2012. Βλέπουμε ότι σε όλες τις ολοκιακές ομάδες το πορτοκαλί αφορά το 2012 η μετάβαση έχει πέσει σε αυτά τα 6 χρόνια. Τώρα όσον αφορά ε, το τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Εξετάσαμε την συζήτηση σχετικά με τις ενιαίες συμβάσεις του χρόνου, το οποίο είναι ενδιαφέρον. Χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία πρότειναν να ε, λήξει ο διεισμός της αγοράς εργασίας, ε, εισάγοντας ένα ενιαίο συμβόλαιο, μια ενιαία σύμβαση, ε, και να υπάρχουν τα ίδια δικαιώματα ε, απόλυσης, όμως ε, έχουν γίνει συζητήσεις πάνω σε αυτό τα τελευταία δέκα χρόνια και στόχος είναι να περιοριστεί το χάσμα μεταξύ των μόνιμων και προσωρινών συμβάσεων και να γίνει μια πιο ισότιμη κατανομή στην αγορά εργασίας, διότι βλέπουμε αυτές τις ανισορροπίες όταν φτάνουμε στο τέλος μια σύμβασης και θα μπορούσε να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο. Δεν έχει υπάρχει αρκετή έρευνα όμως γι' αυτό και επειδή έχουμε δει τις συνέπειες ε, στην εργασία ε, υπάρχουν ακόμα βεβαιότητες πάνω σε αυτό. Ίσως να μην μπορείτε να το δείτε ξεκάθαρα γιατί είναι μικρό στη διαφάνεια, όμως εδώ έχουμε τα διάφορα είδη ε, ε, ενιαίων συμβάσεων που υπάρχουν. Ε, από την μία έχουμε την προστασία στην απόλυση, εάν είναι μεγάλη ή μικρή προστασία και στον οριζόντιο άξονα έχουμε ανησυχία για όλους ή αν διαφοροποιείται ανάλογα με την παλαιότητα ε, στην υπηρεσία και έτσι έχουμε τέσσερα διαφορετικά είδη ε, πάνω αριστερά έχουμε ένα συμβόλαιο λοιπόν το οποίο δεν έχει προστασία από την απόλυση και ε, ισχύει για όλους σε αντίθεση, κάτω αριστερά έχουμε ένα, μια σύμβαση που έχει καλή προστασία από την απόλυση και εφαρμόζεται ε, σε όλους. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο καταργούμε τα, τις προσωρινές συμβάσεις. Οπότε διαφοροποιείται από την άλλη ε, στα, πάνω, ε, στα πάνω δεξιά ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας με, αυτό το, με αυτή τη διαφοροποιημένη σύμβαση λοιπόν που ε, σχετίζεται με την προστασία ε, όσον αφορά την ε, παλαιότητα. Βλέπουμε δηλαδή την ευελιξία που υπάρχει εδώ πέρα και το πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν θα επικεντρωθώ πολύ σε αυτή τη διαφάνεια διότι είναι περίπλοκη. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι ουσιαστικά δείχνει ε, τα, τις δυνατότητες που προφέρουν οι συγκεκριμένες συμβάσεις σε σχέση με το δικό σύστημα. Ε, αν, κατανομή, ε, αν η κατανομή είναι ισότιμη κατά τα πρώτα χρόνια τότε η ε, πολλοί μπορεί να θελήσουν, εργοδότες να θελήσουν να απολύσουν κόσμο πριν γίνουν πολύ ε, κοστοβόροι. Ε, όμως σε ένα διοικό σύστημα έχουμε την επικεντρώση των απολύσεων στο τέλος ε, της σύμβασης και όταν έχουμε σύμβαση λόγω απόλυσης ζήτησης, ε, λόγω απολύας της ζήτησης, ε, αύξησης κόστους, οικονομικών προβλημάτων, τότε πιο πιθανό είναι να απολυθεί κόσμος σε αυτό το πλαίσιο, ενώ σε ένα διοικό σύστημα είναι πιο πιθανό να απολύσουν κόσμο που έχουν ε, μόνιμες συμβάσεις ε, στα στις ενιαίες συμβάσεις είναι πιο, είναι πιο πιθανό να έχουμε περισσότερες προσλήψεις ε, και ταυτόχρονα να αυξηθεί η απασχολησιμότητα με βάση την προϋπηρεσία οπότε έχουμε περισσότερες διακυμάνσεις πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης έχετε μεγάλες ε, διαφορές όσον αφορά τους ε, ετούντες, ε, διότι διαφοροποιείται η κατάσταση ανάλογα με την αποσχολησιμότητα. Βλέπετε λοιπόν και τις χώρες αυτές που έχουμε, 8 χώρες, για να δούμε λοιπόν τι έχουν κάνει αυτές οι χώρες τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασία. Στο πρώτο σημείο, οπότε βλέπετε υπάρχει το ρυθμιστικό πλαίκιο σε ό,τι αφορά τις σχετικές οδηγίες για την ε, προσωρινή εργασία. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια να μειωθεί η προστασία σε ό,τι αφορά τα θέματα απόλυση και δεν αυτά και στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Έχουμε επίση ε, ζητήματα σε ό,τι αφορά ε, πολλές πτυχές της προστασίας από την απόλυση και από την άλλη έχουμε επιδοτήσεις για την ε, πρόθεση των συμβάσεων αυτών όπως στη Σλοβενία και στην Ιταλία. Έχουμε επίση ε, περιορισμού στην ε, διάρκεια των ε, συμβάσεων ορισμένη διάρκεια με, πολύ ευέλικτα όρια και στην Ολλανδία και στην Πολωνία. Σε ό,τι αφορά επίσης την κάλυψη από τα επιδόματα ανεργία, υπήρξε απόπειρα επέκταση αυτών προκειμένου να κινείται ο, ο κόσμο πιο εύκολα μεταξύ θέσεων επασχόλησης και σύντομων ε, τέτοιων ε, συμβάσεων. Κάποια συμπεράσματα. Τώρα επιτρέψτε μου. Οι μεταρρυθμίσει στην αγορά εργασία έχουν κάποιε επιδράσει στην ε, αγορά εργασία, αλλά είναι πραγματικά πολύ αμφίβολο κατά πόσον αυτό έχει μόνιμα αποτελέσματα. Χρησιμοποιούνται αρκετά ευρέω στι πιο πολλέ αγορές εργασίας λόγω της αντίληψης που επικρατεί στους ε, εργοδότες ε, θεωρούν ότι οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις ε, κοστίζουν πολύ και προτιμάνε πιο μάλλον συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αυτή η διτότητα στην αγορά εργασίας αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το επιλύσουμε πολιτικά σε όλες τις χώρες που αποτέλεσαν αντικείμενο της μελότης και δεν έχει εντοπιστεί ακόμα ένα βέλτιστο, ένα ιδανικό μοντέλο για την μείωση αυτής της ζητότητας. Μια τελευταία διαφάνεια σε ό,τι αφορά την απόπειρα ε, εκ νέου ρύθμισης των ε, συμβάσεων ορισμένης διάρκειας προκειμένου να είναι πιο ακριβή, αν θέλετε, αυτή η προσωρινή μορφή απασχόλησης. Είναι πολύ φθηνή στην παρούσα φάση να υπάρχει καλύτερη εφαρμογή και επικοινωνία σε σχέση με τους εφιστάμενους κανόνες. Η... Μεγαλύτερες επενδύσεις στον δημόσιο τομέα και φυσικά χρειάζεται και πιο πολύ έρευνα τομέα σε αυτός γιατί πραγματικά δεν έχει δοθεί επαρκή προσοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και η πρόεδρο, δεν έχουμε μείνει και πολύ γιατί είχαμε μία από τι πιο δύσκολε ψηφοφορίες ε, της ε, θητείας. Ε. Είναι εξαντλημένοι λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι, αλλά ίσως κάποιος θα ήθελε να θέσει ένα ερώτημα. Ναι, η κυρία Γιασλοβιέσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε ότι τα άτομα που έχουν τέτοια σύμβαση ορισμένου χρόνου σπανίως μεταβαίνουν, κάνουν τη μετάβαση σε μια πιο ασφαλή εργασιακή σύμβαση. Σπανίω δηλαδή έχουν μια σύμβαση αορίστου χρόνου. Γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τι δεξιότητε, για παράδειγμα την κατάρτιση των ατόμων αυτών, υπάρχει κάποια έλλειψη ενδιαφέροντο, υπάρχουν ε, ε, έλλειψη, για παράδειγμα, μέσων ε, περαιτέρω κατάρτιση των ατόμων αυτών, προκειμένου να μπορούν να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε συμβάσει αορίστου του χρόνου. Μία ερώτηση ακόμα από τον κύριο Πυρίνσκι να ακούσουμε. Ναι, να κάνω την ερώτησή μου παρά αυτά. Mm. Uh, Έχει να κάνει με κάποια από τα τελευταία συμπεράσματα. Αναφερθήκατε και στην Ευρωπαϊκή Αρχή εργασία που μόλι ψηφίσαμε. Είπατε ότι η καλύτερη επικοινωνία και η καλύτερη επιβολή των νόμων και ενδυνάμωση των επιθεωρήσεων, των έρχων επιθεώρησης. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι κάποιες από τις αρχές επιθεώρησης ε, σε κάποιες χώρες δεν είναι ακριβώς νόμιμες. Yes, Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Για την πρώτη ερώτηση, νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με την ακαμψία της αγοράς εργασίας παρά με τη βούληση των ατόμων. Γενικά από την έρευνα προκύπτει ότι περισσότεροι θέλουν ε, πιο μόνιμη εργασία. Υπάρχουν ε, άνθρωποι που ε, είναι κατάλληλοι και τους ταιριάζει το να έχουν ορισμένου χρόνου συμβόλαια γιατί ανταποκρίνεται στις επιλογές τους αλλά οι περισσότεροι προτιμούν ε, πιο μόνιμες μορφές εργασίας. Δεν είναι ότι δεν θέλουν δηλαδή, απλώς έχει να κάνει με το κόστος ε, της απόλυσης και το γενικότερο κόστος για τις συμβάσεις οριστού χρόνου είναι πιο υψηλά. Έτσι λοιπόν φοβούνται οι εργοδότες ότι δεν θα μπορούν να απολύσουν ανθρώπους που δεν τους κάνουν ή θα είναι πιο ακριβή για αυτούς. Έτσι λοιπόν έχει να κάνει με το σύστημα και την ακαμψία της αγοράς εργασίας. Βέβαια δεν είναι σε όλες τις χώρες δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κάποιες πιο ευέλικτες από όλες, αλλά είναι η εσωτερική δυναμική. Όταν είσαι εντό με μία μόνιμη σύμβαση, σύμβαση του χρόνου, θέλουν οι άνθρωποι να μείνουν, γιατί αυτό είναι λιγότερο επισφαλές. Όμως ε, φυσικά ε, αυτό αποκλείει κάποιους εργαζομένους, ε, αφορά οπότε την δυναμική της αγοράς εργασίας. Και για να απαντήσω στη δική σας ερώτηση, δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν παράνομες πρακτικές. Παραδείγματο χάρη, συμβάσει ορισμένου χρόνου καλύπτουν ε, διάφορε πρακτικέ. Παραδείγματο χάρη, σε ό,τι αφορά την απόσπαση των εργαζομένων, ξέρω ότι έχουμε μια νέα οδηγία και αυτό αφορά την επιβολή. Απλώς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κανονισμοί που υπάρχουν επιβάλλονται και εφαρμόζονται όπως πρέπει. Και φυσικά να ξέρουν και οι εργαζόμενοι τα δικαιώματά τους, γιατί πολλές φορές δεν τα γνωρίζουν κυρίως ε, οι μετανάστες ε, που μεταβαίνουν σε άλλε χώρες και δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα που έχουν. Είναι ένα θέμα τη επιβολής ε, των ε, επιθεωρήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σε εγκαταλείπουν τώρα οι διερμηνείς. Είχαμε ένα δύσκολο πρωινό εδώ στην Επιτροπή. Είχαμε μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις ψηφοφοριών για χρόνια. Είναι εξαντλημένοι λοιπόν οι άνθρωποι. Ευχαριστώ τους διερμηνείς για τη βοήθειά τους και θα ήθελα να σας ευχαριστώ και σε εσά που ήρθατε. Φυσικά παρακολουθούμε το έργο σας και ενημερωνόμαστε για το τι κάνετε, αλλά είναι τόσο απλές αυτές οι διαφάνειες που δείξατε και θα χαιρόμουν αν μπορείτε να μας τις διαβιβάσετε για να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε και εμείς όταν προσπαθούμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους πολίτες στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας εδώ. People are exhausted. But thank you for being here and we are looking forward to to keep in touch with you because you are really dealing with the issues that are on our agenda and in our hearts, I'd say.